της ε, εκτίμησης αντικτύπου. Και βεβαίως αυτό μετά την υιοθέτηση του ψηφίσματος αυτού. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρέντινγκ. Τελειώσαμε τη συζήτηση. Αύριο στις 12 θα γίνει η ψηφοφορία. Ζητώ συγγνώμη για την σύγχυση που επικράτησε. Δεν λειτουργεί εδώ σωστά το σύστημα. Η επόμενη έκθεση είναι η έκθεση Φάλμπερ. Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων πρόκειται για την έκθεση σχετικά με την εξωτερική διάσταση κοινωνικής πολιτικής, την προαγωγή των εργασιακών κοινωνικών προτάσεων και την ευρωπαϊκή εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ελπίζω όλα να πάνε καλά αυτή τη φορά. Για μία ακόμη φορά λοιπόν κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, όπως ήδη σας είπα, στην προηγούμενη παρουσίασή μου, πριν από μερικά λεπτά, η εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής θα πρέπει να προάγει εργασιακές, τα εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα και σε τρίτες χώρες. Η στρατηγική της Σαββόνας και οι στόχοι της Ευρώπης 2020 τονίζουν και προωθούν την κοινωνική διάσταση περισσότερο τώρα από ό,τι παλιά αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ανταγωνιστικότητας και τις διάφορες οικονομικές πτυχές. Γι' αυτό στην έκθεσή μου ε, επικρίνω διάφορα στοιχεία. Αν θέλουμε οι τρίτε χώρε με τι οποίε διαπραγματευόμαστε διάφορε συμφωνίε και συνάπτουμε συμβάσεις, αν θέλουμε αυτέ οι τρίτε χώρε να σέβονται τι αρχέ και, ευρωπαϊκά το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο πρέπει να εφαρμόζουμε αυτές τις αξίες και εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να τις κηρύσουμε. Εάν θέλουμε οι χώρες με τις οποίες διαπραγματευόμαστε συμφωνίες και συμβάσεις να συμμορφώνονται και να τιμούν αυτές τις συμφωνίες, θα πρέπει να σεβόμαστε εμείς αυτούς τους όρους που θέτουμε. Και είναι σαφές ότι παρουσιάζουμε σε πολλές χώρες μας ε, τα διάφορα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εργασίας, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Όσον αφορά ε, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, αυτή σίγουρα είναι μια πολύ καλή ιδέα και ξεκινήσαμε να συζητάμε αυτή την ιδέα την αρχή της δεκαετίας του 70. Όμως, αυτή η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο απαιτούμε και να το επιβάλλουμε. Ακούσαμε να λέγεται ότι έπρεπε να υπάρχει κάποια οδηγία που να καλύπτει αυτά τα θέματα, διότι κάποιες εταιρείες δεν συμπεριφέρονται με έναν τρόπο ε, που δείχνει ότι σέβονται την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Έλαβα πάνω από 150 τροπολογίες Προσπάθησα να τις λάβω υπόψη και θα προσπαθήσω, αλλά εξακολουθώ να επικρίνω διάφορες πτυχές. Θα πρέπει να υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, διότι είναι παράλογο να ισχυριζόμαστε ότι σεβόμαστε τις διατάξεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και να συνομιλούμε με διάφορες χώρες που δεν σέβονται τις αρχές αυτές. Πέρσι συζητούσαμε την οδηγία για το ωράριο εργασίας και ήταν αντίθετα τα μέτρα με την πρώτη συμφωνία που είχε εγκριθεί στο Διεθνή Οργανισμό Εργασίας το 1919. Εκεί τονιζόταν ότι έπρεπε η εβδομάδα να είναι 48 ώρες. Και χαίρομαι που περίφθη αυτή η οδηγία στο Κοινοβούλιο. Αυτά είχα να πω. Δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω. Όλοι γνωρίζετε τα θέματα αυτά. Θα ήθελα να προωθήσουμε την αξιοπρέπεια, τα κοινωνικά δικαιώματα, να σεβόμαστε αυτά που διδάσκουμε τους άλλους, να τα εφαρμόζουμε. Και όλα αυτά, αν τα εφαρμόσουμε τελικά, θα είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Μπασέσκου έχει το λόγο. Εγώ θα να μιλήσω για την άλλη έκθεση όμως, όχι για αυτήν. Um Ωραία. Η κυρία Ντάντσιλα για αυτή την έκθεση. Κύριε Πρόεδρε, οι ευρωπαϊκές στατιστικές έχουν καταδείξει ότι πάνω από το μισό των εργαζομένων στην Ένωση και συγκεκριμένα οι μετανάστες δεν έχουν κοινωνική πρόνοια. Άρα θα πρέπει να έχουμε κάποιο κοινά πρότυπα για μια κοινωνική πρόνοια υπέρ των εργαζομένων. Επίσης κοινέ κυρώσεις για όλους όσους δεν καλύπτουν με τι αντίστοιχε εισφορέ του εργαζομένου του. επόμενο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρέπει να γίνει εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και θα πρέπει να διευκολυνθούν τα αναγκαία βήματα. Επίση, θα πρέπει να έχουμε μια αυθεντική πολιτική δέσμευση των κρατών μελών, ούτω ώστε τα κοινωνικά δικαιώματα να προωθηθούν και οι αντίστοιχοι μηχανισμοί στην Ένωση. Τα κοινωνικά δικαιώματα, αυτά τα οποία κατηχρώνονται από τη συνθήκη θα πρέπει παντού να γίνονται σεβαστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ντάντσιλα. Στανό. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια κύριε Πρόεδρε. Οπότε να σας πω τη θέση μας. Πρώτα πρώτα. Ελπίζω θα χτενίσουμε, θα βελτιώσουμε το τελικό κείμενο πριν τη ψηφοφορία και θα είναι αρκετά δυναμικό, αποφασιστικό για να τονίσουμε το ρόλο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας που θα πρέπει να αναβαθμιστεί. Όπω συμφωνήσαμε και με τον εισηγητή. Εκουσία, εταιρική, ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντική. Όμω, τα κράτη πρέπει τον πρώτο λόγο και οι διεθνεί φορεί δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να μην έχουμε πρότυπα δεσμευτικά όσον αφορά την εταιρική ευθύνη ιδέα και παραβίαση των θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων. Δεν είναι δυνατόν να το επικαλεστεί κανείς ως συγκριτικό πλεονέκτημα. Άρα, να επιμείνουμε σε διμερείς και πολυμερείς σχέσεις με τους εταίρους μας και τα συμπεφωνημένα να τηρηθούν. Ευχαριστούμε κυρία Στανόφα. Και τώρα έχει το ρόλο η κυρία Φιγκερέντο. Ευχαριστώ. Η σύμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας του 2010 αναφέρει Φέρει ότι 20% των εργαζομένων δεν έχουν επαρκή κοινωνική κάλυψη και ότι δεν έχουν κοινωνική ευθύνη οι εταιρείε απέναντί τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται συμφωνίες ελευθερω εμπορίου με αυτές τις χώρες. Το 20% αυτών των χωρών που δεν έχουν κοινωνική ε, πρόνοια χωρίς να απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση οι εργαζόμενοι αυτών των χωρών να έχουν το δικαίωμα για για συλλογικέ συμβάσει και να συνάπτουν συλλογικέ συμβάσει με του εργοδότε, ούτε ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να μην γίνεται διάκριση όσον αφορά την απασχόληση στι χώρε. Και κάλυψη όσον αφορά τα επικίνδυνα επαγγέλματα και απαγόρευση τη εργασία παιδιών. Σε αυτό το 20% των χωρών που δεν έχουν επαρκή μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. Δεν είναι καθόλου ικανοποιητική αυτή η κατάσταση και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να βελτιώσει την όλη κατάσταση. Ευχαριστώ κύριο Πάσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Αληθεύει ότι ακόμα και εντός της ευρωπαϊκή Ενώσεως η κοινωνική προστασία των εργαζομένων πολύ συχνά δεν ε, παρέχει επαρκή κάλυψη. Κυρίως όσον αφορά τους μετανάστες. Ε, εκείνους που θέλ, πρέπει να πάνε σε άλλη χώρα για να βρουν δουλειά, δεν ξέρουν τη γλώσσα, δεν ξέρουν την νομοθεσία της χώρας και πολύ συχνά οι μετανάστες είναι σε δυσχερή θέση εν συγκρίση με τους ντόπιου εργαζομένους. Όμως εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσει να εξασφαλίσει το ότι οι κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας να ισχύουν στις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται με τρίτες χώρες. Γνωρίζοντας την αγορά εργασίας στην Ασία, την Αφρική και άλλες περιοχές του κόσμου, πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι η κατάσταση των εργαζομένων και σε αυτές τις περιοχές του κόσμου θα βελτιωθεί σημαντικά και γι' αυτό προσωπικά υποστηρίζω τις προτάσεις ε, του εισηγητή και πιστεύω ότι ανοίγει ένας δρόμος για τη βελτίωση των κανόνων και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πάσκα. Η κυρία Τικάου. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί θεωρώ πραγματικά ότι όλες οι εταιρείες, όλες οι επιχειρήσεις όπου και αν βρίσκονται θα πρέπει να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η Ευρώπη έχει σαν αποστολή να προωθήσει και να εξάγει το ευρωπαϊκό μοντέλο. Και λυπούμαστε πολύ γιατί δεν υπάρχει μια ομοιογενής ρήτρα έτσι ώστε να μπορούμε να την προτείνουμε σε κάθε διμερή συμφωνία που διαπραγματευόμαστε. Υπήρξε μια οριζόντια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά. Πρόκειται για μια εξαιρετικά φιλόδοξη συμφωνία, μια από τις πιο φιλόδοξες που έχει ποτέ υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σε αυτή τη συμφωνία δεν υπάρχει κοινωνική ρήτρα. Οι δύο χώρες βεβαίως θα το συζητήσουν το θέμα αυτό στο μέλλον. Αλλά λυπούμε πολύ γιατί δεν υπάρχει μια μειογενής δυνατότητα να μπει αυτή η ρήτρα σε όλες τις διμερείς συμφωνίες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τίκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαίρω την Φάμπερ για την κάλυψη των θεοδιαγραφών για το εργατικό δυναμικό στην έκθεσή του και την κάλυψη στο συγκεκριμένο θέμα τη εταιρική κοινωνική ευθύνη. Σήμερα αυτό μα δίνει τη δυνατότητα να επηρεάσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την ανακοίνωση θα προβεί το θέμα και ζητώντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα απ' όλα να κρατήσει ανοιχτό ορισμό όσον αφορά την εταιρική ευθύνη που υιοθετήθηκε στο φόρουμ των πολλαπλών φορέων και να υπάρξει και στι διάφορε εθελοντικέ πρωτοβουλίε να υπάρξει σύγκληση και στι ιδιωτικέ συμφωνίε που ήταν η πρώτερη πολιτική να γίνουν συγκεκριμένε ε, προτάσει για να εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο αυτά οι διατάξει σύμφωνα με τον ΩΣΑ όσον αφορά ε, την εταιρική ευθύνη και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένη χρηματοστατική, περιβαλλοντική κοινωνική αναφορά, συμμόρφωση με όλες τις σφαιρική ε, συμμόρφωση των εταιριών με τις διάφορες αυτές πτυχές. Και θα πρέπει να προωθηθεί η ευθύνη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στον κόσμο και να καλυφθούν οι διαφορές διακυβέρνησης που ε, διαπιστώθηκαν στη μελέτη του Δημβούργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε να σας ε, βοηθήσει, ελπίζω η συζήτηση αυτή να σα βοηθά απόψε κυρία Ρέντινγκ όσον αφορά τι απόψει που εκφράστηκαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χάουιτ. Τελειώσαμε με την διαδικασία Καστριά και τώρα θα δώσω όμως το λόγο στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Ρέντινγκ. Πρόεδρε, εξ ονόματος του συναδέλφου Κλάς Λοάντο, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μας γιατί το θέμα αυτό καλύπτει πολύ σημαντικές πτυχές της κοινωνικής μας πολιτικής και της εξωτερικής της διάστασης. Στηρίζουμε λοιπόν σαν Επιτροπή αυτού του είδους την πρόθεση των προτύπων σαφώς με οικονομικές πτυχές. Στηρίζουμε τη συνέχιση των συζητήσεων, το συντανισμό των προσπαθειών στα πλαίσια του G20, προετοιμασία του G20 για την απασχόληση. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παράδειγμα της μεγαλύτερης συνοχής που προετοιμάζεται παγκοσμίω. Επίση, η Επιτροπή στηρίζει μια στενότερη συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς και μεταξύ διεθνών οργανισμών, ΟΣΑ, Διεθνούς Οργανισμού εργασία, κάτι που είναι καθοριστικό για να μπορέσουμε να παίξουμε ένα ρόλο σε διεθνές επίπεδο και να φτάσουμε σε κάποια διεθνή πρότυπα μια μέρα. Η συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και έχει σαν επίκεντρο μια νέα σύμβαση για τον Διεθνή Οργανισμό Εργασία για τους εργαζόμενους, την κοινωνική προστασία. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αφορά ιδιαίτερα την φετινή συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Τα πρότυπα που εμπεριέχει αυτή η σύμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας θα αποτελέσουν το επίκεντρο των εργασιών. Το σημερινό ψήφισμα υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει αυτά τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας όπως ε, μια πολιτική χωρίς διακρίσεις για την ισότητα των φύλων η Επιτροπή θα συνεχίσει να προωθεί αρχές όπως την αξιοπρεπή εργασία, τα πρότυπα εργασία, την κοινωνική ευθύνη, την βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς όπως η ανάπτυξη και οι εμπορικές συναλλαγές. Το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνεται να παρουσιάσει μία δήλωση, μία ανακοίνωση για την κοινωνική ευθύνη έτσι ώστε να προτείνει διεθνή συνεργασία πρόθεση της αρχής της κοινωνικής ευθύνης με άλλες χώρες με τις οποίες έχουμε συνάψει συμφωνίες. Σκοπός μας είναι να μιλήσουμε για τους νέους, την απασχόληση των νέων, την κατάρτιση, την πολυμορφία, την αναδιάρθρωση, την τοπική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σήμερα εν ώψη των δυσκολιών των οικονομιών που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρέντινγκ. Τελειώσαμε με το θέμα αυτό και αύριο στις 12 θα γίνει η ψηφοφορία. Το επόμενο θέμα είναι έκθεση Μίτσελ για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης για